και από τις 15 έως τις 17 με την ημερήσια διάταξη η οποία έχει δημοσιευτεί στο έγγραφο συνόδου και που φέρει τον ίδιο τίτλο καθώς και στο ίντρανετ.